Τώρα, περνάμε στην ε, τελευταία έκθεση, στην ημερήσια διάταξη. Νικολάη, μετανάστες που διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, η κυρία Νικολάη, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι ανέχεια και η έλλειψη νομικού πλαισίου έχουν οδηγήσει σε ένα μεταναστευτικό κύμα και έχουν θέσει σε βάλωτη κατάσταση ε, τους μετανάστες αλλά κυρίως ε, τις μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα έχουμε μια πραγματικότητα ιδιαίτερα και πιο δύσκολη δεδομένη της οικονομικής κρίσης. Και αν αγνοήσουμε αυτή την ευάλωτη κατάσταση σημαίνει ότι θα ανεκτούμε ένα είδος σύγχρονης δουλείας και αυτό είναι απαράδεκτο για το χώρο ελευθερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες ε, σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους όταν μιλάμε για γυναίκες που δεν έχουν επίσημα έγγραφα και βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κίνδυνη είναι πολλαπλοί και καταρχήν έχουν να κάνουν ε, με την έλλειψη ασφάλειας δικαίου στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες αυτές. Επίσης, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην υγεία ε, δεν τηρείται για τις γυναίκες αυτές. Πολλές φορές οι μετανάστριες δεν έχουν πρόσβαση στην βασική εκπαίδευση στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης ζητήσαμε τα κράτη-μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την Σύμβαση 29 για την καταναγκαστική εργασία. Επίσης, δεν γίνονται σεβαστά σε πολλά κρατη κράτη-μέλη τα εργατικά δικαιώματα αυτών των γυναικών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, έχουν ε, παρουσιάσει την κατάσταση των γυναικών αυτών. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια ηθική υποχρέωση απέναντι στις ε, γυναίκες αυτές, δηλαδή να θέσουμε σε εφαρμογή την οδηγία που έχουμε στη διάθεσή μας και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία. Το πράττω αυτό και στην έκθεση. Αναφέρομαι στην οδηγία για την άδεια παραμονής, την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων που αποτελεί πρόοδο σε νομικό επίπεδο καθώς τα δικαιώματα των θυμάτων ε, δεν σχετίζονται, δηλαδή η προστασία των δικαιώματων των θυμάτων δεν σχετίζεται με την νομική τους κατάσταση. Πρέπει στα κράτη-μέλη να βρεθούν τρόποι να ενθαρρυνθούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό. Οι γυναίκες που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή ταυτόχρονα βιώνουν και τον κοινωνικό αποκλεισμό και θα έπρεπε ως Ευρωπαίοι να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανέχεια και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε στο περιθώριο αυτόν τον πληθυσμό. Έχουμε εκπονήσει κάποιες συστάσεις βάσει των ευρωπαϊκών ιδογιών και βάσει εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και βάσει επιστημονικών ερευνών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ακόμη και αν δεν έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τα άτομα που βρίσκονται σε αυτή την ευάλωτη κατάσταση, θα πρέπει να βρούμε λύσεις για να προσδιορίσουμε ποια είναι τα άτομα αυτά. Σε πολλά κράτη-μέλη, οι μετανάστριες δέχονται πολύ μεγάλες διακρίσεις. Δεν μπορούμε να ενεχόμαστε λοιπόν το φαινόμενο αυτό στην Ευρώπη. Θέλω λοιπόν να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου και ελπίζω ότι η Κομισιόν θα βασίσει στην έκθεσή μου για να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες αυτές. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έδωσε τόση μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό. Αυτό αποτελεί την απόδειξη ότι υποστηρίζουμε τη δημοκρατία και υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γέννη. Ευχαριστώ. Για το ΚΑΤΣΔΙ, η κυρία Μπασέσκου. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Χαιρετίζω την έκθεση της κυρίας ε, ε, Νικολάη και για σήμερα για πρώτη φορά αυτή η συζήτηση για το τι γίνεται με αυτές τις μεταναστές χωρίς έγγραφο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν απολαβούν δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή επικράτεια και όπως αναφέρει και η έκθεση αντιμετωπίζουν διπλή δυσμενή διάκριση και όσον αφορά το καθεστώς που τις διέπει και όσον αφορά το φύλλο τους. Θύματα των δικτύων ε, πορνείας, ε, οργανωμένου εγκλήματος κλπ. Είναι η πιο ευάλωτη κατηγορία της κοινωνίας από κάθε άποψη. Δεν μπορούν να πάνε στις αστυνομίες να βοήθεια. ούτε σε νοσοκομείο δεν μπορούν να πάνε ακριβώ λόγω της νομικής τους θέση. Άρα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, κάποια έτσι, βασική γιατρική βοήθεια και κάποια δικαιώματα στη δουλειά για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Νταντσίλα, παρακαλώ, συνάδελφο Νταντσίλα. Κυρία Πρόεδρε, μία μετανάστρια χωρίς έγγραφα δεν μπορεί να διαμείνει μονίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χειρότερα από έναν οποιοδήποτε κάτοικο τρίτης χώρας. Έχει διπλή διάκριση και λόγω φύλου και λόγω της ε, νομικής κατάστασης και ε, επομένως θα πρέπει κάτι να γίνει για αυτές τις γυναίκες που τους ε, αρνούνται υπηρεσίες υγείας, ε, στέγασης, ε, παιδείας και συνέχεια εφίστανται κακοποίηση ψυχολογική ή σωματική. Αυτοί που καταστέλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτούς ανήκει η ευθύνη. Θα πρέπει να υπερασπιστούν τα δικαιώματα ανηκει η ευθυνη θα πρεπει να υπαρξουν τα δικαιωματα αυτων των μεταναστών, κυρίως των μεταναστριών. Να εφαρμόσουμε το κοινωτικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, γιατί έχει υπογράψει συγκεκριμένε συνθήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια προς την συγκίτρια. Πρόεδρε, είναι σημαντικό να δούμε πόσο μεγάλη σημασία δίνει η έκθεση σε μετανάστριες ε, χωρίς έγγραφα. Αντί λοιπόν να περιθωριοποιούνται οι γυναίκες αυτές, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης στην πηγή. Δηλαδή ε, στις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτές οι γυναίκες. Και να λύσουμε και το πρόβλημα των γυναικών που βρίσκονται ήδη εδώ. Να αντιμετωπίσουμε το θέμα της υγείας τους, της παιδείας τους ε, αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει οι γυναίκες περισσότερες να έρθουν. Πρέπει να προσαρμόσουμε την ε, πολιτική μας και να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθουν μετανάστες, είτε είναι νόμοι είτε παράνομοι. Επίσης, οφείλουμε να μιλάμε για γυναίκες ε, που είναι ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurostat μας λέει ότι το 61% των θυμάτων της ε, εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι περισσότεροι εξ αυτών γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφος Μορβάη, παρακαλώ. Πρόεδρε, Η τρίτη σύσταση της έκθεσης αναφέρει ότι το θέμα αυτό είναι κοινή ευθύνη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Ε, εγώ δεν νομίζω όμως ότι σκεί κάτι τέτοιο και δεν θα υπερψηφίσω την έκθεση. Οι χώρες που είχαν ε, μεγάλες απικίες ε, και εξακολουθούν να είναι πλούσιες χώρες φέρνουν τελείως διαφορετική ευθύνη από ας πούμε τις ε, φτωχές ε, πρώην κομμουνιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, παραδείγματο χάρη από την Ουγγαρία, η οποία τώρα είναι θύμα του νεοπαικιοκρατισμού. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ασχολείται με τις ε, γυναίκες μετανάστες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από φτωχές χώρες που είναι θύματα παράνομης εμπορίας ανθρώπων και άλλων μορφών καταχρήσεων. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, κυρία Νικολά, για την εκθέση αυτή. Μας Επενθυμίζει ότι πολλές μετανάστρες συχνά βρίσκονται σε μία ευάλωτη κατάσταση και μπορούν ε, να υφίστανται διακρίσεις ε, και λόγω του νομικού καθεστώτος και λόγω του φίλου τους. Πρέπει να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση και να δούμε όλους όσους θίγονται από τις δράσεις μας, κυρίως τους πλέον ευάλωτους ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων ε, και των ομάδων όπως ε, των μεταναστριών χωρίς επίσημα έγγραφα πρέπει να διασφαλιστεί και να ληφθεί υπόψη στην εφαρμογή όλων των τυχών της μεταναστοπολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να αντιμεταπίσουμε το πρόβλημα χρειάζεται διεθνής προσπάθεια, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει εδώ να επιστρατεύσουμε και το Διεθνή Οργάνωση Εργασίας θα πρέπει να παρακολουθούμε τη σωστή εφαρμογή των ε, νομοθετημάτων και η Κομισιόν έτσι μπορεί να δυσφελίσει ότι οι μετανάστριες ε, χωρίς εγγραφά ωφελούνται από τις εγγυήσεις που παρέχει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπό την οδηγία επιβολής κυρώσεων στους εργοδότες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα τιμωρούνται όσοι απασχολούν ε, μετανάστες χωρίς έγγραφα στη μαύρη αγορά. Η οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να δέχονται ανώνυμες καταγγελίες. Το μέλλον του 2014 η Κομισιόν θα παρουσιάσει μία έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας τρία χρόνια μετά την προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων για τα κράτη-μέλη. Τώρα δεν έχουμε σχέδια να θεωρήσουμε την οδηγία. Στην έκθεσή σας για την ταχεία και σωστή εφαρμογή ε, αναφέρονται κάποια στοιχεία τα οποία τα καλωσορίζει η Κομισιόν και, ε, θα, έχει ξεκινήσει και η προσπάθεια της μεταφοράς ε, του δικαίου για το ε, λαθρεμπόριο και θα μπορούσαμε στο μέλλον να ξεκαθαρίσουμε τις διάφορες διατάξεις. Η Κομισιόν θα υιοθετήσει το καλοκαίρι μία ανακοίνωση και την πρώτη έκθεση εφαρμογής για την οδηγία περί επιστροφής. Η Κομισιόν θα προωθήσει την αξιοπρεπή μεταχείριση των ατόμων που επιστρέφονται, καθώς και συστηματικές εναλλακτικέ στην κράτηση. Επίσης, συμφωνούμε επί της ανάγκης να επικεντρωθούμε περισσότερο ε, σε κάποιες ε, πρακτικές που να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη σύλληψη και επίσης να ακολουθήσουμε και την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρέπει να παρακολουθήσουμε τη σωστή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και δεν έχουμε άμεσες προθέσεις να προτείνουμε νομοθετικές αλλαγές. Όμως, μακροπρόθεσμα, δεν αποκλείουμε κάποιες ε, τροποποιήσεις. Και τέλος, ε, σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων, να τονίσω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση το εμπόριο ανθρώπων είναι απαράδεκτο και πιστεύω ότι το πολιτικό και νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του εισεμπορίας ανθρώπων λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου του προβλήματος. Και η οδηγία του 2011 για την εμπορία ανθρώπων και η συμπληρωματική στρατηγική του 2012 αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν τη διάσταση του φύλου της εμπορίας ανθρώπων ταυτόχρονα καθώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις συγκεκριμένες πτυχές ε, της διάστασης του φύλου, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δράστες που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους ε, θα μπουν στη φυλακή. Αυτοί αξίζουν τιμωρία και όχι τα θύματα, ενώ δυστυχώς ε, πολύ συχνά τα θύματα αντιμετωπίζονται ως μικροεγκληματίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30. Και η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα αύριο, 4 Φεβρουαρίου 2014. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί και μπορείτε να τη βρείτε στο, στην ιστοσελίδα.